Okay, can you take your seats, please? Για καθίστε. We have a long voting session, so... Η ψηφοφορία θα είναι μακρά.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 Μπορεί να μα ξεφύγει τίποτα και να είναι τίποτα συναρπαστικό. Δεν ξέρει ποτέ κανεί. Λοιπόν, μια που κάθεστε ακόμα και υπάρχει μια κάποια χλαπαταγή, βάλτε τις ε, κάρτες ε, ψηφοφορίας ε, στην αντίστοιχη σχισμή να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες, κάνουμε δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Όποιος προτιμούσε να είναι σπίτι, παρακαλώ να ψηφίσει ναι. Come on, I've got 40 cards plugged in. 40 συνάδελφοι έχουν βάλει τις κάρτες, 35 ψηφίζουν, 37 ψηφίζουν, 38, 39. Δύο δεν έχουν ακόμα πατήσει το κουμπάκι. Right, 42 plugged in and 40... 42. Ένας δεν έχει πατήσει ακόμα το κουμπί. Πάντα ανησυχώ για αυτόν που είναι εδώ πέρα και δεν πατάει το κουμπί. Μήπως είναι κάποιος που νομίζει ότι το έχει πατήσει και δεν πατιέται τελικά. Πέρας της ε, ψηφοφορίας. Okay, so 32 people would rather be at home. Και οι 32, 32 λοιπόν θα προσπαθούσαν να, θα προτιμούσαν συγχωρείτε να είναι σπίτι τους. May I suggest that you send somebody to get one? Αν είναι και δεν έχετε την κάρτα σας, στείλτε κάποιον να τη φέρει. Ναι, εντωμεταξύ θα σας μετρήσουμε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 Okay, right. Now, I'm going to open the meeting. We're meeting start. Λοιπόν, θα ξεκινήσει τώρα η συνεδρίαση. Λίγη ισχύα, παρακαλώ. Ε, δεν θέλω να φωνάζω. Δεν θα ξεκινήσει η συνεδρίαση μέχρι να κάνετε ισχύα. I'm not starting till I have quiet. There's still a lot of noise. Εξακολουθώ να ακούω θόρυβο. There's still a lot of noise. Please. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, συνεχίζονται ακόμα οι συζητήσεις. Θα αρχίσω να λέω ονόματα σε λίγο. Δεν θα ξεκινήσουμε μέχρι να έχουμε ησυχία. I feel like a teacher trying to wait for ε, σαν δασκάλα καμιά, καμιά φορά. βλέπετε, οι γονείς πώς καταλαβαίνουν. Λοιπόν, να εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Ελίσσα έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο για να ζητήσω ακόμη μια φορά και επισήμως την αναβολή της ε, ψηφοφορίας ε, που προβλέπεται σήμερα για το διπλό αυτό πακέτο. Για, και αυτό για δύο λόγους. Όταν το Νοέμβριο μας είχαν δώσει την πρόταση της Κομισιόν, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι τώρα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία πάλι προς την κατεύθυνση της λιτότητας και της πειθαρχία και η πολιτική μας ομάδα πάντα προσπαθούσε να συμπεριλάβει στοιχεία ανάπτυξης και σύγκλησης που δεν υπάρχουν. Το Συμβούλιο μεταστρέφεται. Υπάρχει μια πρώτη συνάντηση μεταξύ Μέρκελ και Ολάντ αύριο, η Γερμανική Βουλή και άνω και κάτω. Άλλαξαν τον χρόνο της συζήτηση για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο Συνόδου Κορυφής. Οπότε δεν μπορεί να συνεχίσουμε να συζητάμε αυτές τις ευαίσθητες λεπτομέρειες όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες γύρω μας. Σας παρακαλώ λοιπόν. Ζητώ την αναβολή της ψηφοφορίας. Δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες από αυτή την αναβολή και ίσως υπάρξουν ε, θετικά αποτελέσματα για την εικόνα και τη δουλειά του Κοινοβουλίου. Η ε, Σας ευχαριστώ. Έχουμε μία πρόταση αναβολής. Κάποιος λοιπόν πρέπει να την υποστηρίξει και κάποιος να μιλήσει κατά αυτής της πρότασης. Θέλει κάποιος να υποστηρίξει αυτή την πρόταση. Ε, προφανώς ακούσαμε ήδη μία ομιλία υπέρ. Σιλβί, εσείς. Δεν θα πω πως ε, συμφωνώ 100% με τους λόγους, αλλά είμαστε υπέρ της αναβολής γιατί θεωρούμε πως το κείμενο δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή και θεωρούμε πως πρέπει να γίνεται καλή δουλειά, σωστή δουλειά στο Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να γίνουν δεκτές και κάποιες από τις ε, τροπολογίες μας. Μάλιστα, κάποιος κατά της αναβολής, Πολ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι κατά της αναβολής για δύο λόγους. Για τους πολιτικούς λόγους ε, που αναφέρει η Ελίζα να πω με όλο το σεβασμό που τρέφω για το πρόσωπό τη, ο κόσμο αλλάζει κάθε μέρα. Ε, και εάν πρόκειται να εξαρτώμαστε από αυτό, καλύτερα στο κατεβάσουμε τα ρολά και α πάμε να κάνουμε του ψαράδε. Ε, γιατί διαφορετικά δεν κάναμε καμιά δουλειά στο κοινοβούλιο. Εγώ νόμιζα πω είμαστε ανεξάρτητοι. Κατά τα λοιπά, κατά πόσο είναι κακή δουλειά όλη αυτή, είναι αυτό προσβλητικό. Γιατί μετά την περασμένη εβδομάδα οι συγητέ και οι σκεώδει συμφώνησαν σε μια πλήρη συμφωνία. Και μόνο στη συνέχεια, επειδή γίναν διάφορε και μυστήριε παρεμβάσει, παρεμβάσεις σε σχέση με τον τρόπο εργασίας του Κοινοβουλίου αρχίσανε να ανακύπτουν ε, θέματα. Γιατί είχαμε βρει συμφωνία για ένα κείμενο που κατά τη γνώμη μας, όλων τη γνώμη, ήταν ε, ε, θεμητό. Γι' αυτό και είμαι κατά της αναβολής. Um, Ευχαριστώ πολύ η ψήφος αυτή να καταγραφεί. Ναι σημαίνει αναβολή, όχι σημαίνει πως συνεχίζουμε με την μερίσια διάταξη ως έχει. Εντάξει. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία επί της αναβολής. Ναι, ίσον αναβολή, όχι, συνεχίζουμε κανονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Voted, Ψήφισαν όλοι, πέρας. And that is, 19 uh, in favor. 19 υπέρ, 21 κατά. Δεν αναβάλλεται η ψηφοφορία. Ωραία. Ελίζα. Um, thank you, Chair. I'll make... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας, ζητώ από τους ε, συναδέλφους και από εσά να δεχτείτε μία αλλαγή στη σειρά των δύο εκθέσεων γιατί είχαμε κάποιες κινήσεις ε, και αλλαγές ε, την τελευταία στιγμή στη δική μου την έκθεση και πρόκειται περί πακέτου. Θεωρώ λοιπόν πως είναι καλύτερο να δούμε πρώτα τη δική μου την έκθεση και μετά τη δεύτερη γιατί στην πρώτη έκθεση έγιναν οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής που μπορεί να θέσουν εν κινδύνο την συμφωνία η οποία είχε επί της αρχής επιτευχθεί και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Γκοζές. Η πρόεδρος, ναι. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα πάλι να ακούσω κάποιον υπέρ και κατά για την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης για να ψηφιστεί πρώτα η έκθεση Φερέρα και μετά η έκθεση Γκοζές. Κάποιος υπέρ? I don't see anybody Udo. Udo. Ναι. Ε, κοιτάξτε, είναι αρκετά περίπλοκα τα πράγματα. Ήδη. Γιατί είδατε και στο παρελθόν πως ακριβώς η κυρία Φερέρα πάντα προσπαθούσε να διατηρήσει μια συνοχή στο κοινοβούλιο και να βρει συμβιβαστικές διατυπώσεις. Και όταν κάνει αυτή την πρόταση και μετά από ένα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το οποίο μόλις είχαμε, το οποίο ήταν ούτως ή άλλως με μικρή διαφορά, νομίζω πως θα πρέπει να την ακούσουμε. Κάποιος άλλος, Ζαν Πολ. Κανείς δεν θα εκλογεί ότι θέλω να ισχύσει η διαδικασία που έχει αποφασιστεί. Έτσι έχει εργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο, οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο τόσο ώστε να αλλάξουν τα πράγματα και δεν καταλαβαίνω ακριβώ τι ωφελεί το να αλλάξει η σειρά. Τι θέλετε, θέλετε να τελείσει ομοιρία το κείμενο ούτω ώστε να αποσπάσει κάποιες ωφελήματα. Τι γίνεται εδώ πέρα, πρόκειται εδώ πέρα για κάποια τεχνάσματα και γι' αυτό εγώ θέλω να τηρηθεί η μερσία διάταξη. Καλά λέει πρόεδρο και τώρα θα ψηφίσουμε. Πι, υπέρ σημαίνει να αλλάξει η σειρά στη μερσία διάταξη. Όχι σημαίνει να μείνουν τα πράγματα όπω είναι. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Δύο δεν έχουν ψηφίσει. Πέρασε ψηφοφορίας. 18-21. Επομένως, η αρχική σειρά πρόβλημα στη διάταξη θα ισχύσει. Και προχωρούμε τώρα στο δεύτερο σημείο. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Σύμφωνα με την διάταξη 73 του κανονισμού μας, σας ενημερώνω ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσει για τα Eurocoins και επομένω έκλεισε σεβασμό με το Συμβούλιο. Επομένω, αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση με την πολιτική μα ομάδα, από τι πολιτικέ ομάδε μάλλον, θα πάει το κείμενο προς έγκριση στη δεύτερη ομιλία του Μαΐου. Υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις. Όχι από ό,τι βλέπω, εμένα σας ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε. Θα με το 3 και 4. Πρόσβαση δραστηριότητα επιστοτικών ιδρυμάτων και προληπτική εκστρατεία πιστοτικών ιδρυμάτων. τα τμήματα 1, 2, 3 του κανονισμού. Έχουμε δύο αλλαγέ. Θα σα πω όταν ε, έρθουμε στο σημείο εκείνο, όταν φτάσουμε εκεί και αν κανεί ε, μπερδευτεί όσον αφορά τη λίστα ψηφορία, να μα το πει. Να αρχίσουμε όμω Ο εισηγητής, ο Ότομαρ Κάρα, θα σα πει δύο λόγια. Ότομαρ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές, τους συνεργάτες μας, τη γραμματεία για αυτά τα οποία έκαναν τις τελευταίες εβδομάδες σε ένα πολύ δύσκολο θέμα με διαφορετικά σημεία που ενδιέφεραν τον καθέναν και παρόλα αυτά καταφέραμε να έχουμε 46 συμβιβαστικές τροπολογίες από τις 163 ε, ε, και σε μεγάλο βαθμό να έχουμε μία συμφωνία. Κάτι το οποίο δείχνει την διάθεση όλων παρά τις διαφορετικές απόψεις να συμβιβαστούν. Και τους ευχαριστώ όλους για τη δουλειά που έκαναν και για τη στήριξη στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Και ξέρω βεβαίως τι σημαίνει αυτό σε ένα τόσο ακανθόδες θέμα, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε και να σταθεροποιήσουμε την τραπεζική αγορά, να υπάρξει ανάπτυξη και να μην υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των τραπεζών. Να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινή γνώμη και να πάμε στις διαπραγματεύσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών. Προσπάθησα να σεβαστώ τις διαφορές δεν ήθελα μόνο πλειοψηφία να έχω. Ελπίζω λοιπόν ο τρόπος ε, με τον οποίο εργαστήκαμε να αποδώσει στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε, Ότμαρ. Επομένως, αρχίζουμε τώρα για την οδηγία. Τροπολογία 78. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καταπίπτει αν δεν εγκριθεί 79, 80 καταπίπτει, 81 και 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 85 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος νομίζω έχει εγκριθεί. Μόνο θα κάνουμε τον έλεγχο. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. Και ε, ε, γκρίνεται 26-17. Νέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92. Υπέρ κατά κατά άποχες έλεγχος για το 90 που νομίζω πάντως ότι εγκρίθηκε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 27, 16 και αυτή εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές και αυτή εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω μπορείτε ότι αλλά κάνουμε έλεγχο. Είναι κάπου διαφορετική εδώ η πλειοψηφία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Καταπίπτει. 22, 22. Ξέρετε, η ισοψηφία τι σημαίνει 108. Υπέρ, κατά, αποχές απολύτωται. Συμβαστική. Ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο συμβαστικό γάμα με προφορική τροπολογία. Και έτσι διορθώνονται παραγραφή 2 και 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πω, από θα τα γινουν Όταν 6-16. 115 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AU. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι και αυτή εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. «126» λέει ο πρόεδρος. Πέρας Δεν Εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψήφισαν όλοι πέρας 22-22 εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές και σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Σηματάφι F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ζήτα G εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, ε, συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται συμβαστική J. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική K. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 164, υπέρ. Κατά. Αποχές. ένοχος για το 164. Ψήφισαν όλοι, πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται 23-22 165 υπέρ κατά αποχές 166 υπέρ κατά αποχές 67 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το πλέον. θα κάνουμε επαλήθευση για το 167. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 23-22. Πλαστική λαμπ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 169. Υπέρ. Κατά. Αποχές. έλεγχος 169 ψήφισαν όλοι απορρίπτεται 20-22 170 υπέρ κατά εποχές 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική μη υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική νη. Υπέρ, κατά, Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. you υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές νομίζω αλλά θα γίνει έλεγχος πέρας εφορίας απορρίπτεται 227 υπέρ κατά αποχές και αυτή απορρίπτεται ρο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 230, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να γίνει έλεγχος. 230. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρας, απορρίπτεται. 22-23. 231 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για το 231 Εγκρίνεται 23-22. Υπέρ. 232. 233 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Δεν οριακή ψηφορία και η πλειοψηφία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 18-27. 234. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά εγκρίνεται 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος 237 ψήφισαν όλοι πέρας Εγκρίνεται 27-18. Συμβαστική S. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 270. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη νέα που δεν καλύπτεται από το συμβασμό. Έχουμε 312. Ψηφίζουμε την 312. Κοιτάξτε τι οδηγίε έχετε. Να σας πω πριν, πρόκειται, πρόκειται για το αίτημα των πρασίνων μέσω της τροπολογίας όσον αφορά τις για το γέννη. Αν θέλετε λοιπόν να προβλέπετε ποσόστοση για το γέννη είναι ναι, αλλιώς είναι όχι. 312 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίτω. 22-22.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 330 in favour. Against. Abstentions. That's rejected. 335 in favour. Against. Abstentions. Can we check 335? Υπέρ κατά. Ε, ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Ένας δεν έχει ψηφίσει ακόμη, πιάσε το ελιτό κομπάκι, κάποιος δεν το έκανε, πέρασε τις ψηφοφορίες τώρα. Καταπίπτει 22-22. Έχει απορριφθεί. Παρακαλώ. Όταν πήρε το κουμπί, να σιγουρεύεσαι ότι έχει ανάψει το φωτάκι. Β. Β. αγγλικό, συμβαστική, που εγκρίνεται. Η 44, Υπέρ, κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική W. να σας εξηγήσω πώς θα ψηφίσουμε για τη συμβαστική αυτή. Ελπίζω έχετε λάβει το κείμενο, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι με άλλη σειρά από αυτήν που μου εξηγούσαν. ψήσουμε τα διαφορετικά κομματάκια που συμμετέχουν αυτή την ε, συμβαστική πρώτα-πρώτα τη ECR ε, και αποτελεί μια προσθήκη για το τέλο και εδώ θα ψηφίσουμε ε, για το καραγόσον θα αναγραφεί 50 ή 75%. Και αν αυτέ απορριφθούν τότε θα ψηφίσουμε το συμβαστικό κείμενο όπω έχει εγκριθεί. Οπότε πρώτα πρώτα η προβολή του τη ECR. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές θα γίνω όμως έλεγχος ψήφισαν όλοι άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν ένας ακόμη δεν έχει ψηφίσει όλοι ψήφισαν 10.35 απορρίπτεται και τώρα θα ψηφίσουμε για το 50%. Ψηφίζουμε. Γίνεται ηλεκτρονικά κατευθείαν για το 50% ψηφίζουμε. Άλλοι δύο, άλλος ένας. Μήπως κάποιος μπάτα κάτω το κουμπάκι πέρασε. Α, 20-24. Και τώρα. Ελεκτρονικά και το 95%. Ψηφίζουμε. Άλλη τρεις, άλλη Όσο μας ψηφίζουμε πέρας, απορρίπτονται και αυτή. Και τώρα, ψηφίζουμε την συμβαστική που, με τη μορφή που είχε προηγουμένως, χωρίς τις μεταβολές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 351. 351. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 351. Άλλοι δύο, άλλος ένας. Πέρασε οφορίας. 23-22. Εγκρίνεται. Συμβαστική Χ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 372. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 373. Υπέρ. Έλεγχος. είναι δικιά μου και γι' αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ελπίζω τα έκανα σωστά, Αλλιώ θα βρω τον πελά μου. A lot more people to vote yet. Ακόμη πολλοί δεν έχουν ψηφίσει. Five more people to vote, four more, three more, two more. Anybody else vote? Κάποιο άλλο θα ψηφίσει, ένα. Πέρα τη πληροφορία. Εγκρίνεται 27 υπέρ 18 κατά. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 374 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y, Y, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ζήτα, υπέρ ναι. κατά αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 385 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 389 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α, α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 395 υπέρ κατά Κάποιοι δεν έχουν ψηφίσει, αλλά να κάνουμε έλεγχο στην 395. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται με 27 υπέρ, 18 κατά, 396 υπέρ. Κατά. Αποχές και αυτή εγκρίνεται 407 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίνεται συμβαστική αβ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 420 υπέρ κατά εγκρίνεται 421, ε, 422, εγκρίνεται 421, 22 και αυτή εγκρίνεται 424 υπέρ. Κατά. Τα αποχές εγκρίνεται 425. Εγκρίνεται 426 υπέρ. Κατά. το αποχές εγκρίνεται 427 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται σε 28 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. AC υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική AD. Βρωκή τροπολογία η οποία αφορά αυτόν τον οδηγό φράκτη. Υπέρ κατά κατά εποχές πρέπει να ψήσετε πρώτα πρώτα την προφορική τροπολογία άρα θα ψηφίσουμε πήραμε μόνο για την διατύπωση της προφορικής τροπολογίας και εγκρίνεται 23-22. Και τώρα παρακαλώ να ψηφίσουμε όσον αφορά την ε, τοπολογία με την προφορική. Υπέρ, κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο 450 υπέρ κατά αποχές πρέπει να Εγκρίνουμε. Άρα καταπίπτει 21-21. 451. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 452. Έλεγχο για το 451. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται 36-9. Άρα Βίκη. Είχα δίκιο. Παρασύρθηκες, παρασύρθηκες, γιατί έχεις πάει καλά πριν. Τελούσα 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος Ψήφισαν όλοι. Πέρας. That's carried. Εγκρίνεται. 25-18. Συμβαστική ΑΕ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική AF ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Okay, compromise AG. AG υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 502. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 502. Ψηφισαν όλοι πέρας και εγκρίνεται 23-22. AH. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 522 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AK, συμβαστική υπέρ μισό λεπτό έχουμε εδώ προφορική τροπολογία να ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία τα Ευκολότερα έτσι. Είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Εγκρίνεται και τώρα η συμβαστική με την προφορική τροπολογία εγκρίνεται. 524 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 525 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 526 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται 527 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AM υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται AV υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 534 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 535 υπέρ κατά 535 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται έλεγχος για 535 Ψηφίζουμε 235 Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 25-18. Άρα η 536 καταπίπτει. AN ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AO ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 552 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε έλεγχο για το 252. ψήψαν όλοι. Ακόμη ένας πέρας. Απορρίπτεται. 21 υπέρ, 23 κατά. 39 υπέρ κατά αποχές 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές α εγκρίνεται η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική IP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να ελέγξουμε το για το 47 ψηφίζουμε τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές έλεγχος δεν μπορώ να διακρίνω τα χέρια τα υψωμένα 48 ψήφισαν όλοι πέρας νομίζω ότι εγκρίνεται εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές 49 έλεγχος Everybody's voted, votes. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. Απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να γίνει έλεγχος γιατί δεν δείχνονται καλά τα χέρια τα ψωμένα Ψήφισαν όλοι. That's Εγκρίνεται. Δεν έχει, δεν έχει πολλές. 51. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 52 και 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται οι δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 55 κατά καταπίπτει, αν λέει, δεν έχει εγκριθεί 103. Τι γίνεται με What? 173 has been adopted. βλέπω ότι έχει εγκριθεί. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε την 55. Πήνα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική A, Q. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ρ, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος επί του 69 Ένας με ψήφισε, πέρας, 27-18 εγκρίνεται. 70, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AT ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε τώρα στο 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές έλεγχος επί το 75 Everybody's voted. Votes closed. Πέσαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται 22 υπέρ 23 κατά. Και τώρα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Four more, three more. Άλλη τέσσερις, άλλη τρεις, ε, κανείς άλλο να ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίες. Πέρας. 43, 43 υπέρ και ένας κατά χωρίς αποχές. Το ψήφισμα για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψήφισαν όλοι. Και άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν πέρας της Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν πέρας τώρα. 42 υπέρ και ένας κατά. Χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Έχουμε πολλή δουλειά μας ακόμα μπροστά μας. Και τώρα θα προχωρήσουμε. Πρώτο τμήμα. Πάμε στη λίστα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 μέρος πρώτο κάντε ησυχία μέρος πρώτο συμβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική β υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.39 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική γ υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Να επαληθεύσουμε την 298. Να Άρχεται η ψηφοφορία. Άλλοι τέσσερις ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Ψήφισαν όλοι. Δύο ακόμη. Πέρας. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 24-18. 2,99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. είπαι. υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές ακτή. Τροπολογία. 3.55 και 3.56 εγκρίθηκαν. Όχι. 3.57 υπέρ. Κατά. Ορίστε. 3.57 κατά. Αποχές απορρίπτονται. 354 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 361 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική κάπα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μάλιστα. Συμβαστική L με προφορική τροπολογία στο τέλος μέσα με πολλαπλά μερίσματα δεν θα επιτρέπονται σε συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 1.3α της οδηγίας. Θέλουμε να ψηφιστεί χωριστά yeah, okay. All those in... υπέρ της προφορικής τροπολογίας κατά αποχές. Φαίνεται πως απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν ψήφιση της συμβαστικής απολογίας χωρίς την ε, προφορική υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά περνάμε στην M υπέρ κατά. Νομίζω πως είναι δεκτή. Γιατί και το L είναι υπέρ, ναι. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 409 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 415 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 άρα νομίζω καταπίπτει ε, κύριο συγητής καταπίπτει την ψηφίζουμε μάλιστα 416 υπέρ υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 417 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική νη υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 422 και λοιπές υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. Να, να την επαληθεύσουμε την 422. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Α, απορριπτεται 1529. 15-29. όμικρον υπέρ κατά αποχές δεκτή. Π υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4.34 με προφορική τροπολογία. Νομίζω αυτές μπορούν να πάνε μαζί υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω πως είναι δεκτή. Να την επαληθεύσουμε. Την 4.34 με την προφορική τροπολογία. Δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Τέσσερις ακόμα. Θα κλείσει η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 28-14. 4-35 πέρα Κατά. Αποχές. Απορρέ... Να επαληθεύσουμε 4 4-35 γιατί κάτι περίεργο γίνεται εδώ πέρα. Ψήφισαν όλοι. Θα κλείσει η ψηφοφορία. Ναι, δεκτή. 4.36 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 4.37 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές δεκτή 4.56 περ κατά αποχές απορρίπτεται 4.60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε την 4.60 Ψήφισαν όλοι, δύο ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Μάλιστα, πέρας. 7 υπέρ, 36 κατά. Δεν ήταν και τόσο μικρή διαφορά. Συμβαστική S. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4,98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4,99 υπέρ αποχές απορρίπτεται. 500 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 501 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 502 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 503 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 504 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τάφ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική για μια στιγμή. Όχι, πάμε πίσω, πάμε πίσω. Υπήρχε μια προφορική τροπολογία στην ΤΑΦΑ, τώρα την είδα. Προφορική τροπολογία λέει Μάλιστα. Αποκατάσταση γυμνασίου. Αυτό ήταν σε περίπτωση που δεν ε, περνούσε. Έγινε δεκτή λοιπόν η συμβιβαστική. Η ΤΑΦ. Περνάμε τώρα στην συμβαστική U. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5-14 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 5-14. Τρεις ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Θα κλείσει την ψηφοφορία. Δύο ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Δεκτή. 26-17. 5-15 υπέρ κατά αποχές 5.16 5-16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5-17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5-18 καλύπτεται οπότε καταπίπτει συμβαστική W υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική X υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή Μάλιστα. Έχουμε την ΑΒ με προφορική τροπολογία των σοσιαλδημοκρατών. Μια αρκετά μακροσκελής και θα ψήσουμε αυτήν πρώτα. Συμβαστική λοιπόν ΑΒ με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Τέσσερις δεν έχουν ψηφίσει. Θα κλείσω την ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, 24 κατά. Περνάμε στην αρχική συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 5.87 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 588 υπέρ κατά Ποιοι είναι κατά παρακαλώ τις 588 να την επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί δεν μπορώ να διακρίνω Τέσσερις δεν έχουν ψηφίσει, τρεις. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 21-20. Και πολλοί δεν ψήφισαν. 589 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική AC υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΑΕ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 600 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 601 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 602 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AF Έχουμε μια προφορική τροπολογία του ECR. Να ψηφίσουμε πρώτα αυτήν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική στο σύνολό της υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 603 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. AG υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 605 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. AH υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. AI υπέρ κατά αποχές δεκτή AJ υπέρ κατά αποχές δεκτή 622 υπέρ κατά αποχές δεκτή AK υπέρ κατά αποχές δεκτή AL υπέρ κατά αποχές δεκτή AM με σοφορία σε δύο μέρη Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε την συμβαστική χωρίς το 16β και μετά το 16β. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο, υπέρ κατά αποχές δεκτό. 639 υπέρ κατά αποχές δεκτή. AN υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προσπαθώ να βρω πόσες είναι οι προφορικές τροπολογίες. Είναι ίδια δύο φορές, μάλιστα. Προφορική τροπολογία του ECR για την έκθεση στεγαστικά δάνεια. Πρώτα προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και συμβαστική σύνολο της υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 9 Όχι, όχι μια στιγμή. Πίσω, συγγνώμη. Βιάστηκα. Συμβαστική AP με προφορική τροπολογία που θα λέει παράγραφος 1 και ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές δεκτή και συμβαστική με αυτή την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα 669 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική AQ σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 696 υπέρ κατά άποχες να επαληθεύσουμε την 696 Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Κάτι θα άλλαξε λοιπόν. AR υπέρ κατά αποχές δεκτή AS σε τρία μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές δεκτή Τώρα πάμε στην 7-16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7-17 που αφορά μόνο το γαλλικό κομμάτι υπέρ κατά αποχές Πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό. Γιατί υπάρχει αλλαγή μόνο στα γαλλικά. Είμαι πάντα περίεργη με αυτά τα πράγματα. Τι, είναι άλλοι κανόνες στη Γαλλία. Ζαν Πολ, για να εξήγα. Αν στα αγγλικά δεν πρόβλημα, αλλά στα αγγλικά, αν θυμάμαι καλά, το πρόβλημα είναι ε, το, το, το πρόβλημα τη ορολογία μεταξύ credit buy και location. Ε, δηλαδή, πρέπει να γίνει εναρμόνιση των όρων των σχετικών με μίσθωση, χρονομίσθωση κλπ. Δεν τα ψηφίζουμε αυτά συνήθω. Όχι, κατά κανόνα όχι. Διόρθωση είναι αυτό. Διόρθωση είναι αυτή, Μάλιστα. Συμβαστική AT υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική AU υπέρ κατά αποχές δεκτή. AV υπέρ κατά αποχές δεκτή. 727 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Ε. Άλλε 4-3, δεν έχουν ψηφίσει, 2 πέρα. Απορρίπτεται. 20 με 22. 7-28 υπέρ, κατά Αποχέ. απορρίπτεται. AW υπέρ, κατά αποδεκτή. 7-37 υπέρ, κατά απόχέ, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά δεκτή 7.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική A6 υπέρ κατά αποχές δεκτή AY υπέρ κατά αποχές δεκτή. AZ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 749 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μάλιστα περνάμε κατευθείαν στο μέρος δεύτερον. Δεν ψηφίζουμε τον κανονισμό μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Έχετε το κομμάτι αυτό, τα χαρτιά αυτά μπροστά σας. Είστε έτοιμοι. Τροπολογία 750 υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 750. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εντάξει. Δεκτή. 56 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. AAA σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Ορίστε. Πρώτο μέρος στις 3α υπέρ κατά αποχές. Μα δεν βλέπω να τους πράσινους. Δεν, δεν ψηφίζεται. Φιλίπ. Πρέπει να επαληθεύσουμε το πρώτο μέρος της 3α. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερο, υπέρ. Κατά. απόχέ, Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 756 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΑΑΒ υπέρ κατά αποχές δεκτή 765 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται AAC ε, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 766 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Μάλιστα να κάνουμε τις 7.67 μέχρι 7.74. ...7.67 με 7.69 τότε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 7.71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7.72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 773 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 774 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά δεκτή IAD υπέρ κατά αποχές δεκτή AAE σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά εποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά εποχές δεκτή AAF υπέρ κατά εποχές δεκτή 791 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 792 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 793 υπέρ κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε την 793. Ψήφισαν όλοι. Δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα. Ψήφισαν. Πέρας. Απορρίπτεται. 7.95 υπέρ. 7.95 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται 798 υπέρ κατά αποχές δεκτή 800 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή 801 υπέρ κατά αποχές δεκτή 802 υπέρ κατά αποχές δεκτή 803 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 804 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 805 υπέρ κατά αποχές δεκτή 806 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 807 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 808 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. AAG υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. AAH υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. AAI υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα περνάμε στο τρίτο μέρος του καταλόγου ψηφοφοριών και και αυτό είναι επίσης σε δύο μέρη. Μάλιστα, είναι όλοι έτοιμοι. 63 υπέρ, 64 υπέρ κατά αποχές δεκτό, 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 8-14 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή δεν, δεν μπορώ άμα δεν βλέπω το 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 816 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 817 υπέρ κατά αποχές δεκτή AAJ ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή AAK ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή AAL ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 8, 28 υπέρ κατά Ε, συγγνώμη, αλλά πρέπει να ψηφίζουν όλες οι ομάδες. Αλλιώ θα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Θα επαληθεύσουμε λοιπόν την 828. Ε, επαλήθευση ηλεκτρονική. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ελπίζω. Επί τις 8.28 ψήφισαν όλοι, πέρας, απορρίπτεται. 829 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 830 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 831 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή 832 υπέρ 8.33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. AAM υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. AAN υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. AAO υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8.56 υπέρ Όπα. Α, προφορική τροπολογία. Μάλιστα, είμαι διόρθωση. 856 λοιπόν προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 859 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 860 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 861 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. AAP υπέρ κατά αποχές δεκτή AAQ υπέρ κατά αποχές δεκτή AAR υπέρ κατά αποχές δεκτή AAS με μία προφορική τροπολογία Α, δούμε πρώτα την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε. Προφορική τροπολογία επί της AAS. Ναι, να κλείσει η ψηφοφορία. Δεκτή, 25 με 17. Οπότε συμβαστική με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Okay. We, we, we love that tune. Ναι, εντάξει, ωραίο το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, επαληθεύουμε την AAT. Συγγνώμη, AAS. Πέντε δεν έχουν ψηφίσει, τέσσερις, πέρας, 38 υπέρ. 2 κατά. AAT ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 891 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 892 υπέρ κατά αποχές δεκτή ABD με προφορική τροπολογία της ΓΚΟΕ. Πρώτα την προφορική τροπολογία της ΓΚΟΕ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβεστική με την προφορική υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8.99 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 900 υπέρ. Συγγνώμη, μα δεν μπορεί να γίνει έτσι ψηφοφορία. 900 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. AAU υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 912 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. AAV υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. AAW υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή AAX με προφορική τροπολογία των πρασίνων που νομίζω πως είναι διόρθωση οπότε θα τα δούμε μαζί υπέρ Ότμαρ θες να ψηφιστεί χωριστά η προφορική τροπολογία μάλιστα θα κάνουμε την προφορική τροπολογία τότε υπέρ κατά αποχές νομίζω πως έγινε δεκτή αλλά να παληθεύσουμε λίγο την προφορική τροπολογία ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή και τώρα ψηφίζουμε για τη συμβιβαστική ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΑΑΙ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 927 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ADF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Okay, there's first of all there is an oral. Καταρχήν υπάρχει μια προφορική τροπολογία για το πρώτο τμήμα και ποιοι είναι υπέρ της προφορικής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η προφορική τώρα ψηφίζουμε για την συμβιβαστική χωρίς ε, κάποια σειρά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και στη συνέχεια ψηφίζουμε για τις συνθήκες CDE, τους όρους CD και E. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα προχωράμε πολύ. Φτάνουμε στη σελίδα 20 στο, μου, στο δικό μου κατάλογο Ψηφοφορία 19 στο δικό μα. συμβιβαστική αβα υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. αββ υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. ABC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ABD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ABE καταρχήν με μια προφορική τροπολογία των πρασίνων. Θα, ακούσουμε, θα ψηφίσουμε πρώτα την προφορική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και η συμβιβαστική μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην ε, ABF με προφορική τροπολογία από το ECR. Πρώτα την ε, προφορική υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται, συμβιβαστική όπως ήταν υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην ε, τροπολογία, τροπολογία ε, 1168. Ποιοι είναι υπέρ. 1168 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ABG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12-18 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την τροπολογία 12-18. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 12-18. Oh, hang on. We've now got one... Μισό λεπτό. Ένας ε, παραπάνω είναι από το ΕΛΚ τώρα. Ένας παραπάνω ψηφίζει από το ΕΛΚ. Κάποιος που μόλις μπήκε να ξαναβγεί από την πρίζα. Come on, I've got to have one EPP. Άντε παιδιά, ένας λιγότερο στο ΕΛΚ να βγάλει την κάρτα του. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2 υπέρ, 23 κατά. Συμβιβαστική ABI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABM with ABM, μια μικρή σύντομη προφορική που λέει θα αποκαλυφθεί στην 1η Πρώτου 2015 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγξτε παρακαλώ, να θα το ελέγξει. προφορική για την συμβαστική ABM, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, προφορική στην ABM. Ένας ακόμα να ψηφίσει. Τέλος της ψηφοφορίας. 26 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική ABM υπέρ. Oh, hang on. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τώρα έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της ABM. Παρακαλώ ησυχία. Ησυχία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ ποιοι είναι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 1264. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. 1264. Voted, votes closed. Τέλος Μάλιστα. Απορρίπτεται 16 υπέρ 27 κατά. 1296, all those in favor, against abstentions rejected. 1296 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1297 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 12.98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12.99 με προφορική τροπολογία του εισηγητή δική μου τροπολογία ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 13.00 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται ABN Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1308, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1309, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1310, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ABO, υπέρ, κατά, αποχές, 1315. 13-15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13-14 υπέρ Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 13-14 παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. ABP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABR υπέρ... Α, όχι, προφορική. Προφορική για την μη εξαίρεση συστημικών εταιριών υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. for more to vote. Okay. Any more for vote? Votes closed. That's carried. 20. Uh, Then compromise ABR with the oral amendment. ABR λοιπόν με την προφορική που εγκρίθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1338 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ABS μάλιστα ABS αποχές εγκρίνεται ABT σε διάφορα τμήματα Okay. You haven't got this in your voting list, so you've got... Το έχετε στον κατάλογο ψηφοφορίας, αλλά όχι ολόκληρο και πρέπει να με ακούσετε προσεκτικά. Please, please, can you... Σας παρακαλώ, ακούστε με λίγο. It's all right. I'm, I'm about to tell you... Θα σας πω τι γίνεται εδώ, λοιπόν. Γιατί είναι κάπως καινούριο. Ούντο. Κοιτάξτε, μια τεχνική ερώτηση για την ομάδα μου. Στον κατάλογο ψηφοφορίας υπήρχε ένα λάθος και θα ήθελα να σας το δείξω. Να σας δείξω, θα σας δείχνω τι θα πρέπει να ψηφίσετε. So, here we... Μάλιστα, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, στην εισαγωγική παράγραφο, δηλαδή χωρίς τις γλώσσες για έκθεση για έκθεση σε έναν ή περισσότερο τομεί περισσότερους τομείς, περιφέρειες ή κράτη-μέλη. Εδώ έχουμε λοιπόν την εισαγωγική παράγραφο χωρίς αυτά τα λόγια. Ε, ποιοι είναι υπέρ. Against. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και εγώ τα έχω χαμένα.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 Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 19 κατά 24 υπέρ. Μετά έχουμε την εισαγωγική παραγραφό 1β. Με τις λέξεις για κάθε έκθεση, για έκθεση σε, σε έναν περισσότερους τομείς. Oh, Κοιτάξτε, είναι πολύ περίπλοκο αυτό που έχω εδώ στον καταλογό μου. Ελπίζω εσείς να έχετε καταλάβει καλύτερα. Τώρα λοιπόν ψηφίζουμε για τις λέξεις που αποκλείσαμε ώστε να ξαναμπούν σε αυτή την παράγραφο που λέει για κάθε έκθεση, για έκθεση σε έναν ή περισσότερους τομείς, περιφέρειες ή κράτη-μέλη. Υπέρ ποιοι είναι, κατά, αποχές, Πρέπει να το ελέγξω. Okay, is everybody voted. Votes closed. That's 21. Τέλος ψηφοφορίας 21 υπέρ, 21 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. We have a, a separate vote. Και τώρα έχουμε χωριστεί άλλο τμήμα ψηφοφορία για τα σημεία Β μέχρι και K στην πρώτη υποπαράγραφο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έπειτα έχουμε τα σημεία K, B μέχρι K, E. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει Πρέπει να ψηφίσουμε για την ABT γιατί την αλλάξαμε.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 Την ψηφίσαμε χωρί τι λέξει τη ε, προφορική που λέει για κάθε έκθεση για έκθεση σε έναν ε, ε, περισσότερο τομεί περιφέρειε ή κρατημέλη. Ζητώ συγγνώμη που ήταν έτσι τόσο περίπλοκη. Και πάμε στην 1360. 1360. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική ABU με προφορική τροπολογία. για την περίφραξη των ε, μικρομεσαίων. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική με αυτές τις λέξεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1384 και οι υπόλοιπες ήδη που είναι ταυτόσιμες κατά, αποχές ε, εγκρίνονται ε, συγγνώμη, απορρίπτεται 1389 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται 1390 υπέρ. 1390. Μπορείτε να μου πείτε τι ψηφίζετε. Υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 1391. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1392 υπέρ κατά 1392 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για τη 1392 voted, votes closed. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 23 ε, υπέρ, 21 κατά. Τι τι, ναι, δεν πιέσατε το κουμπάκι. Ωραία, 23 προς 22. Εγκρίνεται και πάλι. What you mean? You voted the wrong way. Okay, look, let's... Ψήφισες λάθος. Αντάξει, άντε, ας ξαναψηφίσουμε για να είμαστε βέβαιοι. 13.92 ψηφίζουμε. Come on. Can everybody vote? There's two more to vote. Ψηφίστε παρακαλώ. Δύο ακόμα κουμπάκια πρέπει να πατηθούν. Δύο, δύο. Τέλος της ψηφοφορίας. Ε, τώρα είναι 21 υπέρ και 22 κατά. Κάποιος ξυβανίστη. Α, δεν... 39... Come on.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 five more, more, more, more. If you push your buttons, it's quicker. Μα άμα πατάτε τα κουμπάκια γρήγορα, τελειώνουμε και γρήγορα. Τέλος της ψηφοφορίας. 26 υπέρ 18 κατά. 13.94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13.95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ABW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1403 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως εγκρίνεται μπορώ να ελέγξω τη 1403 ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 1403 Voted, votes closed. Τέλος της Τώρα έχουμε έναν παραπάνω ΕΛΚ. Ωραία, τέλος της Εγκρίνεται. 30 υπέρ, 12 κατά. Come on, we've got Άντε παιδιά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Πάμε στην επόμενη. ABX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14-23 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ελέγχουμε. Three more to vote. Τρεις ακόμα. Τέλος ψηφοφορίας. Καταπίπτει. 22-22. Συμβαστική ABY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ABZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ACD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ACE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ACF καταρχήν την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1462 υπέρ κατά αποχές mm-hmm. απορρίπτεται. ACG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1471 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1476 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ACJ τώρα ψηφίζουμε για αυτήν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ACK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1482 υπέρ κατά αποχές Βίκυ, Δεκατέσσερα είμαστε. Λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 1482. Ε, it will be open. Everybody's voted, votes closed. That's... Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 27 προς 18. ACL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. That's ACM. Uh, ACN. ACN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15.04 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15.05 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ACP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μάλιστα Τώρα έχουμε τις δύο εναλλακτικέ για το αν θα Έχουμε να ψηφίσουμε για την εναλλακτική 1, που σημαίνει ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω νομοθεσία. Η εναλλακτική 2 ε, είναι η κατεξουδότηση πράξη. Αν θέλετε την κατεξουδότηση πράξη, θα ψηφίσετε όχι στην εναλλακτική 1. Λοιπόν, συμβαστική ACQ, εναλλακτική 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εναλλακτική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Compromise ACE. Πάμε στη συμβαστική ACR. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ACS. Έχουμε και εδώ δύο εναλλακτικέ. Η πρώτη είναι η νομοθεσία και η δεύτερη είναι η κατεξιοδότηση πράξη. Πρώτα, εναλλακτική 1 λοιπόν, η νομοθεσία υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Εναλλακτική 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην συμβιβαστική ACT. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1596 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1597 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ACV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ACW με προφορική τροπολογία. Πρώτα ψηφίσμα για την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική με την προφορική λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16-13 υπέρ κατά να ελέγξουμε για την 16-13 και την 16-14. 13 και 14 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται 22 προς 20. Συμβιβαστική ACX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, ACZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16-17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16-18 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται 16-19 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ 16-19 voted? Votes closing. Votes closed. That's 16-20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1621 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ADA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16-30 Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1631 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το επόμενο κομμάτι είχε αποσυρθεί και πάμε στην 1637 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1638 υπέρ. Λοιπόν, αν μπλοκ από τη 1638 μέχρι 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Sorry, Ramon. Πάμε τώρα στα εκτιμώντας. 140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 Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ, κα, υπέρ κατά Ας το ελέγξουμε αυτό 154 και 155 ελέγχουμε Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κα, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 165, δεν σηκώνετε τα χέρια σας. So, one too many e Ένας παραπανήσιος ΕΛΚ. Να βγει από την πρίζα. All right, votes closed. That's 21 in υπέρ, 24 κατά. amendment 3 in against abstention. 163 υπέρ κατά αποχές. η 3 ήταν, συγγνώμη. Εγκρίνεται. 167 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά, κατά. Κοιτάξτε, άμα έχω δύο ομάδες που δεν ψηφίζουν δεν μπορώ να προχωρήσω. Εκτονική ψηφοφορία για την 168. Has every voted? Votes closed. Well. 169 in favour, against abstentions carried. Ε, γκρίνεται 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Και πάμε στην... Uh, first part, all those in favor, again. Πρώτο τμήμα λοιπόν, υπέρ, ναι. ναι θέλω... Για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Ψηφίσαμε την αιτιολογική 48. Το α εις 2 την εδώ και κατόπιν ψηφίζουμε την 48β αιτιολογική παράγραφο. Ορθώς και αυτό το λέω γιατί θέλω να σας επισημάνω ότι πρόκειται για παραπάνω από δύο ψηφορίες. Α, καλά λέει πρόεδρος. Οπότε έχουμε το πρώτο μισό του 48α και μετά έχουμε το δεύτερο ήμιση αυτό το οποίο μας ετονίσατε έχετε δίκιο και μετά το υπόλοιπο ανάλογα με το τι θα περισσέψει. Το πρώτο τμήμα πι είναι υπέρ, πι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται και κατά το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. We check the second part. voted. Ψήφισαν όλοι. Ναι. Α, πάλι έχουν ψηφίσει παραπάνω έλκα από ό,τι πρέπει. Καλώς. Τόσο, πέρας εγκρίνεται 25-19. Και τώρα το υπόλοιπο της ειδολογικής παραγράφου είναι υπέρ. Against. Abstentions, that's carried. αποχές, εγκρίνεται. Now we go to amendment 172. 172 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 ε, 179 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές oh, work this. 181. <clears throat> 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Απορρίπτεται, απορρίπτεται, λέει η πρόεδρος. Επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, α, δέλτα, δέλτα, με προφορική τροπολογία προωθήσουμε την προφορική. Πρώτα. Π είναι υπέρ της προφορικής για το ADD, α, δέλτα, δέλτα. Κατά αποχές, α, οριακή πλειοψηφία. Ας γίνει ηλεκτρονική παρήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Και τώρα η υπόλοιπη συμβαστική ΑΔΔ υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. A, D, G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Έλεγχος. 207. 207 by Pavance and Liam, I think. Has every voted? Votes closed. That's 26 to 8. Οριακή αποτέλεσμα 26-18. Favor. Against abstentions. Μας κατά αποχές εγκρίνεται 208, 209 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 210 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές να γίνει έλεγχος για το 2 12 Ψήφισαν όλοι υπέρ ψηφοφορία, εγκρίνεται με 23 ή 21 ψήφου. 2-13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 και 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2-16 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2-19 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2-20 υπέρ κατά αποχές αποχές δεν ξέρω 2-20 έλεγχος voted, votes closed. Πέρα τη οφορίας. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 221. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για το 224 We're checking 224. Έλεγχος του 224. Πέρασε ο χωρίος. Εγκρίνεται. 25-18 και τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Άλλοι τρεις. Πολύ ωραία. Πέρας. 44. 0-0. Right, one more, one more on the legislative resolution. Άλλη μια ψηφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. I nearly I keep forgetting to vote myself every now and then. Come on, there's 11 more to do. Μόνο άλλα 11 μένουν. Παρακαλώ, βρείτε, βρείτε, βρείτε ενέργεια για το νομοθετικό ψήφισμα. Παρακαλώ, λέει πρόεδρο. Συνεχίστε, συνεχίστε. Άλλοι 5, άλλοι 4. More to vote, two more. Two more to vote. 5, 4, 3, 2, ένας λέει πρόεδρος για να ψήσουν ακόμα, άλλο ένα για να πατήσει το κουμπάκι. One too many EPP. <laughs> Και τώρα ψήφισε ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Any EPP. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Εμπρό λοιπόν, βγάλτε τον από την πρίζα. Πέρασε. 44, 0, 0. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, σας προτείνω ένα time out λίγων λεπτών. Okay, we're taking, we're taking a five minute break. Πεντάλεπτο, πεντάλεπτο time out, λέει ο Πρόεδρος. Okay. Okay, can you sit down and I can... Για καθίστε για να, για να δω εάν επιστρέψατε όλοι, λέει ο πρόεδρος. Ah oui, oui, bien sûr. One day. As not in the middle after the vote. Okay, I mean, that's fine. It's your decision, you're the chair. It's not It's not usual, but, no. but it's not prohibited, so it's, it's discretion. I, I don't think. Okay. Please, if you could take your seats, because we. Καθίστε αν θέλετε, διότι. Διότι έχουμε και άλλες ψηφοφορίες. Είπαμε ότι έγινε ψηφορία για το προηγούμενο θέμα της δημοσιονομικής εποπτείας και τη χρηματοδομική σταθερότητα και τώρα θα είπαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις ε, διαμετές με το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού. Η Επιτροπή μας θα αποφασίσει σε σχέση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Θέλετε κάτι να πείτε? Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για το αποτέλεσμα αυτό το οποίο ενίσχυσε τη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου, αυτό είναι αναμφισβήτητο, πέραν από τις ε, συμβαστικές προτάσεις και σας παρακαλώ να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν συντομότερον οι διαπραγματεύσεις. Είναι έτοιμο το Κοινοβούλιο, ελπίζω να είναι και το Συμβούλιο. Thank Σας ευχαριστούμε. Όπως προβλέπουν οι διαδικασίες, η διαπραγματευτική εντολή θα είναι η έκθεση την οποία μόλις εγκρίναμε. Και η διαπραγματευτική ομάδα θα είναι η πρόεδρος, οι εισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές. Και θα σας ενημερώνουμε ως συνήθως συντονιστές, επιτροπή και τα λοιπά. Να σας πω επίσης πως ο πρώτος διάλογος για την ε, οδηγία ε, κεφαλαϊκών απαιτήσεων είναι 13 Μαΐου. 30 Μαΐου, με συγχωρείτε. Η Κομισιόν είναι εδώ πέρα και θέλει να μιλήσει, αλλά δυστυχώς έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Οπότε θα... Εντάξει. Μας ευχαρίσει η Κομισιόν, τελείωσε, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Συγγνώμη Μάριο, γιατί μετά θα θέλει να μιλάει συνέχεια η Κομισιόν και δεν θέλω τώρα να ανοίξω αυτό το κουτί ακόμα και για τόσο σημαντικό θέμα. Ξέρουμε πως ήθελες να μας ευχαριστήσεις. Οπότε τώρα περνάμε στην ε, ψηφοφορία για την έκθεση Γκοζές. Να μιλήσω. Όχι, λέει η πρόεδρος. Εντάξει, θεωρούμε ότι μας ευχαρίστησες. Αλλά στις 8 η ώρα θα σβήσουν τα φώτα στην αίθουσα και έχουμε εδώ πέρα ε, πολλά πράγματα να κάνουμε. Έκθεση Γκοζές. Είμαστε έτοιμοι. Ελίζα, θες να μιλήσεις. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γκοζές και τους συγητές για τη συνεργασία και ήθελα επίσης να κάνω, να πεθύνω μία παράκληση. Η σοσιαλδημοκράτες κατά λάθο δεν αναφέρεται ότι υποστηρίζουν όλες τις συμβαστικές, αλλά τις υποστηρίζουν όλες, πλην της AA και AN, όπου υπάρχει ψήφος κατά συνείδηση. Τις υπόλοιπες τις ε, στηρίζουμε όλες, από δικό μου λάθος δεν αναφέρεται αυτό στον κατάλογο. Μάλιστα, σοσιαλιστές λοιπόν, πλην αυτών των δύο, τις στηρίζουν όλες. Ζαν Πολ, περνάμε στην ψηφοφορία. Ωραία. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική β. Δεν δεν Να επαληθεύσω. Δεν Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε την 8. Ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, κάποιος είναι παραπάνω από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, πέρας. 25 υπέρ 18 κατά. 92 καταπίπτει. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και τώρα που πάμε 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική ή e, υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική A υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται J υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστικές κάπα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές δεκτή. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική εν υπέρ κατά αποχές δεκτή. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ναι. Συμβαστική R κατά αποχές δεκτή. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική τάφ υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική γιού υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική ΒΙ υπέρ κατά αποχές δεκτή 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική W υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική X υπέρ κατά αποχές δεκτή Y υπέρ κατά αποχές δεκτή Z υπέρ κατά αποχές Δεκτή. AA υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. AB υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. AC υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Διακόσια υπέρ κατά αποχές δεκτή. AD υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΑΕ υπέρ κατά αποχές δεκτή 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 να την επαληθεύσουμε. Ψη... Πέρας. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε γιατί δεν βλέπω εδώ πέρα κανένα πράσινο. Ε, ξέρετε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές δεκτή. AF ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 208 υπέρ κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Ένας ακόμα δεν έχει ψηφίσει. Ευχαριστώ. Ψήφισαν όλοι. Δεκτή. 23 με 20. 2-10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2-12 υπέρ. Κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε. Πέρας. απορρίπτεται. 2.11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. AG υπέρ κατά αποχές δεκτή. AH υπέρ κατά αποχές δεκτή. AI υπέρ κατά αποχές δεκτή. AJ υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.20 υπέρ κατά αποχές δεκτή AL υπέρ κατά αποχές δεκτή AM υπέρ κατά αποχές δεκτή AN υπέρ Α, προφορική τροπολογία Πρώτα αυτή θα ψηφίσουμε υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. AN όπως ήταν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Θα Δεν Επαληθεύω την AN. Έχουν ψηφίσει ακόμα δύο, ένας. Πέρας, ευχαριστώ. Δεκτή, 25 με 17. 2,29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 2.33 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται α υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. AP ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Να την επαληθεύσουμε όμως θέλετε. 2.44. Γιατί κάποιοι οπωσδήποτε δεν ψήφισαν. Δύο ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Δεκτή. AR ε, repair. Κατά αποχές δεκτή. Ε, AS υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.47 υπέρ είναι ταυτόσιμη μάλιστα 2.48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.53 υπέρ κατά αποχές δεκτή AW υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 τη απασχόληση υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, AX υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, AY υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή AZ ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 69 Πέρας. Δεκτή. 70 υπέρ. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή επίσης. AAA υπέρ κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 και λοιπές υπέρ κατά αποχές δεχτεί. 79 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 79. Πέρας. Απορρίπτεται για τα καλά. 80 υπέρ κατά αποχές απορριπτεται αβ υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 83 υπέρ ο εισηγητή εδώ πέρα έχει σημειώσει πλήν. Δεν, δεν μ' αρέσει αυτό που λέει ο κύριο εισηγητά. 83. Μην, μην μπείτε μετά. Λοιπόν, 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μάλιστα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του κειμένου όπω τροποποιήθηκε. Δύο ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Ένας ακόμη, πέρας. 25 υπέρ, 4 κατά 13 αποχές. Τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. 13. Και τώρα θα ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα. 4. Δεν έχουν ψηφίσει 2, Ένας. Ψήφισαν όλοι. 26 υπέρ. 3 κατά 14 αποχές. Ναι. Κάποιες μετακινήσεις είχαμε. Να εξηγήσω λίγο σύντομα την ψηφοφορία. Εμείς ήμασταν υπέρ των συμβαστικών τροπολογιών. Οι αποχές που είχα συστήσει ήταν ακριβώς επειδή ήμασταν στο διπλό πακέτο και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τίποτα. Ελπίζουμε να υπάρξει κάποια βελτίωση To the outside world. Και μια πιο έτσι, επικαιροποίηση των μηνυμάτων που στέλνουμε προς τα έξω. Yes, right, okay. Right, okay. Πρόεδρος. Πού? Α, είναι επόμενη. Okay. You Yeah. Oh, okay. Right. Yeah, I keep it. here. Off, off we go. Um, this is now for the. Και τώρα έχουμε την έκθεση. Φερέρα. Τροπολογία 47. Ποιο είναι υπέρ. Τροπολογία Φεραίρα. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Α, είναι ταυτόσημε. Επομένω πάμε 49. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική. Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Βαστική Β περκατά κατά αποχές εγκρίνεται. Σ Περκατά κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος 131 Άλλοι δύο, άλλο ένα να ψηφίσει πέρα. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική Δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ε. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 169. Υπέρ 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, εδώ έχουμε μία κατά ψηφοφορία σε τρία σημεία για το G. G. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα πολύ πιο κάτω. Πάμε στο 209 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 232 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Ι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνονται. συμβαστική J υπέρ αυτή, αυτή είναι σημαντική η γραμματεία J, J, ποιο είναι υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά πρέπει να κάνουμε έλεγχο για το J Everybody's voted, votes closed. Εγκρίνεται. 27, 14. Συμβαστική κάπα, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Λάμδα, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μη, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Νη, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. να και 43 καταπίπτουν διότι έχουν καλυφθεί. Όμικρον. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 274. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 275. Καταπίπτει, καταπίπτει και πάμε 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλω να κάνω έλεγχο για το 276 έλεγχος ηλεκτρονικός για την 276 Right, vote's closed. That's rejected, so... Απορρίπτεται, το 276. Προφορική τροπολογία ε, στην, ε, ε, στην συμβαστική π. Πρώτα η προφορική. Υπέρ, κατά, αποχες εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία όπως τροποποιήθηκε, υπέρ, κατά, αποχές και εγκρίνεται. 283, uh, all in 283 υπέρ κατά άποχες ένα ε, έλεγχος για το 283 283 ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται 22-20 284 κατέπεσε 285 υπέρ 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 285 αν θέλετε να κάνουμε επαλήθευση ψηφίζουμε το 285 Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Άλλος ένας. Πέρασε. και εγκρίνεται 2018. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. μόνο ένα απασχόλησης 1, 2, 3 ένα-δύο συγγνώμη αποχέ εγκρίνεται. Ε, ρο υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική ρο α υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική σίγμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά. Γίνει ελεγχός έλεγχο για το 77. 57, συγγνώμη, για το 57. 57. Closed. Εγκρίνεται. Επασχόληση υπαριθμών 3 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Επασχόληση 4 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΤΑΦ υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά εποχέ, Εγκρίνεται. Οι επόμενες δύο καταπίπτουν των πρασίνων. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινώνται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική U υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινώνται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινώνται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική V. Γκρίντιν. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική W. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για την 83. Okay, we've had some wrong voting, so we'll check 83. Κάποιοι ψήφισαν λάθος, οπότε θα γίνει για το 83. Το είδα, το είδα το χέρι σας, το είχατε σηκώσει. To vote. Πέρασε. Εγκρίνεται. 27. Άρα Κατά τα βλέπω. Χ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87. Έλεγχος. Το ψηφίζουν αντίθετα. Εγκρίνεται. 20-21. Συμβαστική ύψιλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την ύψιλον. Όχι, όχι, εντάξει, εγκρίνεται. Ζήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α. Α, υπέρ, κατά. Συμβαστική ζ α, υπέρ. Ζ α, υπέρ. Υπέρ, κατά. Α, αποχές, εγκρίνεται. Είναι πολύ δύσκολο ο Ζων Πολ να κάνει και τα νοήματα όταν το μιλάνε. 98 υπέρ. 98 υπέρ κατά αποχές που να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλφα αλφα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλφα β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. AC, ε, ΑΣ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 105 Έλεγχος για το AC. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 27-17. 105 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτονται 107 υπέρ κατά εποχές απορρίπτονται 108 υπέρ κατά εποχές απορρίπτονται 109 υπέρ κατά εποχές απορρίπτονται 110 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτονται. AD υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ελεκτρονική κέντρο ψηφορία στον αυτό το σύνολο του κειμένου όπω τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. Και ένα, ναι. 18, 12 και 14 εποχές. Και ψηφίζουμε τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Το οποίο και πρέπει να ψηφίσετε. Άλλοι 11 που δεν ψήφισαν πέντε, 3, 2. και άλλος ένας πρέπει να ψηφίσει. Πέρα ψηφοφορία. 20 υπέρ, 11 κατά και 13 αποχές. Μην φεύγετε, δεν μπορείτε να φύγετε, δεν πρέπει να φύγετε, διότι θα πρέπει να συζητήσουμε και τα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Γκοζές. Αν μου επιτρέπετε, έχω κάποιες παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε. Οι εργασίες και η ζήμωση για αυτό το, στις δύο εκθέσεις έγιναν με τον πιο ορθό τρόπο σε πνεύμα συνεργασίας. Και την προηγούμενη εβδομάδα καταλήξαμε σε συμφωνία εισηγητού και σκιωδών των βασικών πολιτικών ομάδων. Διαπιστώνω ότι μόλις έληξε αυτή η διαδρομή αντίθετα με το τι ισχύει στο Κοινοβούλιο και το νέο αυτό που λέω αντίθετα με το τι ισχύει στο Κοινοβούλιο οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων παρενέβησαν και με διάφορες χειραγωγήσεις προσπάθησαν να ανατρέψουν τη συμφωνία των εισηγητών και σκιωδών. Δεν αξίζει το κοινοβούλιο τέτοιου είδου ε, κινήσει. Όταν μια επιτροπή δουλεύει και ε, ε, έχει έτοιμο ένα θέμα, δεν θα πρέπει να, να υφίσταται τέτοια μεταχείριση. Τέτοιε χειραγωγέ. Η πρόεδρο. Φεραίρα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους ε, εισηγητές και σκιωρές που ενευλάγησαν στο έργο αυτό. Ήταν ε, με, με ανοιχτό πνεύμα και όπως είπαμε και στην αρχή η ζωή συνεχίζεται. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε ένα πάρα πολύ δυναμικό μήνυμα. We are sending Δυνατό μήνυμα, έλεγα, προς την Ολομέλεια και προς ε, τους διαπραγματευτές. θα πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι δεν ήρθε τώρα η κρίσιμη στιγμή, τόσο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μόνο με μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Γι' αυτό το Κοινοβουλίο θα πρέπει σοβαρό το τρόπο να εμπλακεί και σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό είναι το μήνυμα μας που θα πάει στην Ολομέλεια για τελική ψηφοφορία και ελπίζουμε ότι τελικά θα μπορέσουμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις στο έργο που ήδη επιτελέστηκε τόσο ώστε να στείλουμε ένα κείμενο το οποίο να είναι πιο κατανοητό. Αυτούς που εκπροσωπούμε, τους Ευρωπαίους. Thank you. We, we are not normally going to enter... Πρόεδρος, δεν προβλέπεται συζήτηση γιατί έχουμε την ε, Μάριον. Και αν μιλήσει ένα, θα μιλήσουν κι άλλοι. That can't be covered by the rapporteurs. I tried to do a declaration in the name of, to explain the vote. Μάριον. Να σε εξηγήσω τις θέσεις πολιτικής ομάδας και θα πω στα Ολλανδικά. Κυρία Πρόεδρε, ο συντονιστής μας εξήγησε πως ε, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά εισηγητής και σκιώδης εισηγητές. Ε, κάναμε κάποιες συμφωνίες τις οποίες, τις οποίες εμείς σεβαστήκαμε. Παρά το ότι 5 και 10 λεπτά πριν από την ψηφοφορία είχαμε αλλαγές και αυτές μας δυσκόλευσαν στο να τις σεβαστούμε. Τα άρθρα στο διατακτικό λέγαμε πως ε, πρέπει να εγκριθούν και τώρα βλέπουμε πως πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο διάσωσης υπό κάποιες συνθήκες και παρόλα αυτά υπερψηφίσαμε. Αλλά να πω το εξής, υπερψηφίσαμε σε ένα πνεύμα συμβιβασμού, ξέρουμε πως πρέπει να διαπραγματευτούμε, αλλά όσον αφορά το Ταμείο Διάσωση και οποιαδήποτε άλλο, άλλη δυνατότητα να υπομισθούν όλοι από κοινού το χρέος, λέμε πως δεν είναι δυνατόν. Μιλάμε για 2.300 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει λοιπόν να πούμε πως είναι μια τελευταία λύση ανάγκης και όχι η πρώτη στην οποία θα πρέπει να καταφεύγουμε. Οπότε βεβαίως θέλουμε να συνεργαστούμε, αλλά ήθελα απλά να ξεκαθαρίσω τη στάση του ΕΛΚ πάνω στο ταμείο αυτό της διάσωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο εάν θα πρέπει να συνεχίσουμε με μια προσπάθεια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Υποθέτω λοιπόν πως οι συγητές ε, οι συγητές ε, ήθιστε να, λαμβάνουν το λόγο για να μιλήσουν για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Ζαν Πολ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ξέρω να κάνω λογαριασμού και έκανα. Η Μαριάν Τάισεν είπε ξεκάθαρα τι, είπε, τι συνέβη. Εγώ είπα τι θεώρησα λυπηρό και έριξε τις ευθύνες σε ορισμένους που υποτίθεται ότι έκαναν ε, επικοινωνία ή ότι βρήκαν τις λύσεις που δεν μπόρεσαν να βρουν. Δεν έχουμε σαφή εδώ για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και άρα θα πάμε σε πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια. Εγώ αυτό προτείνω. Δεν ξαναρχίσουμε ατέρμονες συζητήσεις. Είτε θα πρέπει ούτως ή άλλως να υποκληθούμε ενώπιον του Συμβουλίου, ε, οπότε δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε ως Κοινοβούλιο, είτε θα πρέπει να προεράσουμε την πρώτη ανάγνωση στον Λομέλια. Η κατάσταση όμως είναι πολύ σοβαρή, κυρίως στην Ελλάδα, και πρέπει να πάψουν αυτά τα παιχνίδια πρωτη αναγνωση στην ολομελεια το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο, που θέτουν, ε, αμφισβητούν τη, τη ζωή και το μέλλον ολόκληρων λαών και νομίζω ότι η ευθύνη μας ε, ε, επιτάσσει να κάνουμε το καθήκον μας. Η Ελίζα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε στον Λομέλη και να ενισχύσουμε την εντολή μας και να την ε, ξεκαθαρίσουμε, να την αποσαφηνίσουμε. Α, μάλιστα. Οπότε, αφού αρχικά η απόφασή μας ήταν να μετακρατήσουμε αυτά ως πακέτο και έχουμε διαφορετικέ απέψει ανάμεσα στου ηγητέ. Εσεί είστε αντίθετοι στην έναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να το ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή. Για το αν δηλαδή τελικά θα ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει για συμφωνία πρώτη. Μήπω δεν κατάλαβα καλά. Ο Ζαν Πολ, ναι, αυτό θέλει. Ah, right, ah, Α, συγγνώμη. Κοιτάξτε, ε, εμείς συμφωνούμε να πάμε στην Ολομέλεια. Το αμέσως. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Ωραία. Πάμε στην Ολομέλεια. Οπότε ο πρώτος τριμερής διάλογος θα γινόταν αύριο, σε 6 δεν θα γίνει λοιπόν. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία, πάμε στην Ολομέλεια. Ναι, εντάξει, το αποφασίσαμε. Ωραία, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, συμφωνούν. Ωραία. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής είναι στις 21 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ, γεια σας. Next week.